ήταν μια καινοτομία, χρειάστηκε να βρούμε την κάποια θέση εκεί. Εν γέννη όμως θα πρέπει να πω πως τα πράγματα εξελίχθηκαν ικανοποιητικά. Ίσως ε, δύο παρατηρήσεις για να κλείσουμε. Να πω ότι η αίσθησή μου είναι ότι αυτό το Ίδρυμα του Τωρίνου, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα δηλαδή για την κατάρτιση, είναι μια μικρή δομή που παίζει όμως ρόλο πολύτιμο όσον αφορά τις συμβουλές που δίνει στις χώρες γιατί έχει μια τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που έχει συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια των ετών και είναι ανεξάρτητη από τους χρηματοδότες. Αν και οι γνωμοδοτήσεις μας λαμβάνονται υπόψη από την Κομισιόν για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αρρωγής, αλλά το γεγονός ότι μπορούμε να εργαζόμαστε ανεξάρτητα από την Παγκόσμια Τράπεζα ή άλλους δωρητές, επέτρεψε στο Ίδρυμά μας, νομίζω, να βρει τη σωστή του θέση χάρη στην εμπειρογνωμοσύνη τους και δεύτερο στοιχείο κλείνοντας, και νομίζω αυτό ήταν και ο στόχο τη μεταρρύθμιση του κανονισμού, το να ανοίξει δηλαδή το πεδίο εφαρμογή τη κατα... της επαγγελματική κατάρτιση από την αυστηρή επαγγελματική κατάρτιση στο πεδίο της, του ανθρωπίνου κεφαλαίου, δηλαδή γενικότερα παιδεία, κατάρτιση, απασχόληση γιατί φυσικά μια κατάρτιση που δεν οδηγεί σε επασχόληση δεν είναι και πολύ χρήσιμη. Μπορεί να είναι μάλλον χρήσιμη από πολιτική άποψη και από άποψη καλλιέργεια, αλλά δεν ε, μπορεί να μα δώσει τα ζήν. Ευχαριστώ κύριο Παλαιοκρεσά. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι σε σχέση με τις συστάσεις που κάνετε για μένα. Είπατε ότι αντικαταστάθηκα Ελπίζω να μην ε, έχουν παρανοήσει τα μέλη της Επιτροπής και να θεωρούν ότι δεν ήμουν αποτελεσματικός και με ε, αντικατέστησαν. Ναι, Ελπίζω. The, the truth is, uh, as you know, Madam Chair, uh, Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, ε, έλαβα την ευγενική προσφορά της Επιτροπής ε, για να ανανεώσω τη θητεία μου, όμως την απέρριψα για σειρά λόγων που δεν θα σχολιάσω εδώ. Uh, Θα ήθελα να σας παραπέμψω ε, στην ε, ε, τρισέλιδη έκθεση ολοκλήρωση της θητείας μου που ελπίζω να διανομηθεί και στα μέλη της Επιτροπής. Σας την έχω ήδη διαβιβάσει. Θα έλεγα λοιπόν ότι η στις σχέσεις μου με, τον, με το Ίδρυμα κατάρτισης έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν άρχισαν οι εξωτερικές αξιολογήσεις από αυτή την Επιτροπή. Βεβαίως και στο παρελθόν είχαν γίνει τέτοιες αξιολογήσεις, αλλά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της χρονικής στιγμής. Συγκεκριμένα άλλαξε η εντολή του ίδιου του Ιδρύματος πριν από τρία χρόνια, όπως ξέρετε, σε μεγάλο βαθμό. και τα συμφραζόμενα σε σχέση με τις ε, παρεμβάσεις ε, του Ιδρύματος ε, στην περιοχή της Βορείου Αφρικής. Έχει αλλάξει η Αρδίνη διότι όπως γνωρίζετε έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει η πολιτική συγκυρία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σχολιάσω τα συμπεράσματα αυτή τη σύντομη έκθεσή μου. Λέμε ότι οι έσκατε εξελίξει στη Νότια Μεσόγειο συνιστούν μεγάλη πρόκληση για το ευρωπαϊκό ίδρυμα κατάρτιση, ώστε το την ικανότητα που έχει να προσαρμόζεται στι νέε εξελίξει. Παρ' όλα αυτά, δημιουργείται έτσι μια μεγάλη ευκαιρία για το ίδρυμα, ώστε να έχει ακόμη πιο προεξάρχοντα ρόλο και επιρροή στην περιοχή και πιστεύουμε ότι τώρα που γίνεται η εξωτερική αξιολόγηση είναι εξαιρετικά ενδεδειγμένη χρονική στιγμή ω προ την εφαρμογή τη εντολή ε, ε, κατά τι εξωτερικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με τι χώρε τη Βορείου Αφρική. Ο μόνο στόχο που δεν μπόρεσε με ξέπιστο τρόπο να καταμετρήσει αυτή η διαδικασία αξιολόγηση είναι η ανάπτυξη ενδογενών ικανοτήτων ε, για την πολιτική επαγγελματική κατάρτιση τόσο στο σχεδιασμό τη όσο και την αναθεώρησή τη και την εφαρμογή τη, διότι πλέον οι Αραβικέ χώρε που μεταβαίνουν στη δημοκρατία αντιμετωπίζουν ζητήματα ζωτικής οικονομικού χαρακτήρα, όπω παραδείγματο χάρη καταπολέμηση τη ανεργία των νέων, ε, προσαρμογή πραγματικέ ανάγκε τη αγορά εργασία ε, ε, και επίση ανάγκε ω προ την ανάπτυξη ανθρωπίνου κεφαλαίου. Συνεπάγονται ανάγκη για υψηλή τεχνική αρρωγή που θα μα δώσει από τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Λειτουργεί ω διεθνή δωρητή, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτιση και έτσι αντιμετωπίζει μια μείζωνα πρόκληση σχετικά με τον νέο σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογή για αυτές τις χώρες. Τέλος, είναι γενικά αποδεκτό ότι καμία αξιολόγηση δεν είναι τέλεια. Ε, το θέμα εγκυρότητα και αξιοπιστία ε, τίθενται ούτω ή άλλω σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό και εξαρτώνται από τη μεθοδολογία και τα, εργαλεία, τα εργαλεία για την έρευνα και για τη συλλογή αυτών των δεδομένων. Δεν συνιστά εξαίρεση η παρούσα αξιολόγηση, όμω οι αξιολογήσει είτε εσωτερικέ είτε εξωτερικέ ε, σε ακόμη πιο χρήσιμο εργαλείο σε αυτή τη συγκυρία που είπαμε συνεπάγεται μεγάλες προκλήσεις για το Ίδρυμα Κατάρτισης, όχι τόσο ως προς το ποιος φέρει τις ευθύνες τελικά κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, αλλά ως προς τα εργαλεία διάγνωσης, ούτω ώστε να προσανατολίσουμε μελλοντικέ πρωτοβουλίες για περαιτέρω βελτίωση του Ιδρύματος, αλλά και κυρίως σε με την αποτελεσματικότητα και τη σημασία των αναγκών των ίδιων των δικαιούχων. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια σε σχέση με το παρελθόν ως προς την οργάνωση και τη σχέση του Ιδρύματος με τις διάφορες διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Σας ευχαριστούμε κυρία Μωρήλ, ευχαριστώ κυρία Σαρτιέ. Σας ευχαριστούμε για την διοργάνωση της σημερινής ακρόασης. Εγώ ε, εξακολουθώ να έχω αμφιβολίες για διάφορα σημεία. Βασίζομαι στα έγγραφα που μας ε, διαβιβάσατε και θα αναφερθώ και στις παρεμβάσεις ε, των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης. Λοιπόν, σημειώνουμε ε, την αποφασιστικότητά σας ε, να αναπτύξετε το ανθρώπινο κεφάλαιο σε αυτές τις χώρες, να προσφέρετε τεχνογνωσία, ώστε να αναβαθμιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα και συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε αυτές τις χώρες. Παρ' όλα αυτά έχω ακόμη κάποιες ε, απορίες. Πρώτον, είδαμε ότι ακολουθείτε ε, την ε, στρατηγική σας, αλλά επί της ουσίας ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής. Στο μίσο που δραστηριοποιείστε, Πώς προλαμβάνετε τα προβλήματα, δηλαδή εάν βασιστούμε σε ένα στιγμιότυπο της κατάστασης, και υπό το φως ε, των στόχων που καλούμαστε να επιτύχουμε μέχρι το 2020, τι κάνετε ε, για την δραστηριοποίηση και την εκπαίδευση των νέων στις χώρες όπου δραστηριοποιείστε, διότι γνωρίζουμε ότι ταυτόχρονα με τις νέες εξελίξεις θα χρειάζονται όλο και περισσότερες δεξιότητες αυτές τις χώρες. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό. Δεύτερον, τι είδους συμβουλές δίνετε για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος των χωρών αυτών. Είδαμε, όπως το είπατε κι εσείς, ότι με την ε, Αραβική Άνοιξη άλλαξε άρνηνη κατάσταση, όμως θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε σχετικά με την κατεύθυνση που θα έπρεπε να πάρει αυτή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στις χώρες αυτές, ώστε να ε, καλύπτονται οι προσδοκίες ε, των λαών, αλλά και να γίνονται σεβαστές οι νέες ισορροπίες που έχουν επιτευχθεί ανάμεσα στις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γειτονικές αυτές χώρες της Νοτίας Μεσογείου. Τρίτη ερώτηση. Τι προκρίνεται για την ενίσχυση τις σχέσεις ανάμεσα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αφενός και την απασχόληση αφετέρου. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μου δώσετε διεξοδικότερες απαντήσεις για αυτά τα τρία ζητήματα. Ευχαριστούμε, κύριο Σέρκας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε ήδη την ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση, τουλάχιστον με τον κύριο Μεζιέρ, που ήταν με ένα πάρα πολύ ενημερωτική και ε, μετά από μια επίσκεψη στο Τουρίνο είχα αποκομίσει και την εξή αντίληψη. Υπάρχει ένα παράδοξο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάρα πολύ χρήσιμο μέσο και εργαλείο, αλλά μου δίνει την εντύπωση και θέλω να ρωτήσω και τους δύο μιλητές μας. Μου δίνει λέω την εντύπωση ότι υποχρησιμοποιείται αυτό το τόσο πολύτιμο εργαλείο. Δεν το αξιοποιούμε όσο θα έπρεπε. Είναι ιστορική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους γείτονές της και τους εταίρους της που θέλουν να συνεργαστούν με εμάς και είναι ε, ιστορικές ε, θεαματικές οι αλλαγές. Έχουμε λοιπόν εμείς ένα μέσο που θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μία από ε, τις ανησυχίες τους και τα μελήματά τους. Πώς θα προετοιμάσουν ε, την νεολαία τους, πώς θα την καταρτήσουν, πώς θα την εκπαιδεύσουν. Μπορεί να είναι σε μια θαυμάσια καταπληκτική Ιταλική πόλη, αλλά είναι μακριά ε, αυτό το Ινστιτούτο και το Ίδρυμα. Έχουμε δυνατότητες, τι οποίες όμως δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα και υποδομές που χρειάζεται. Το... Ρωτώ, βέβαια, εκείνο που συνεχίζει έχει κάποια σύνεση, αλλά ο Ποχωρών θα μπορούσε να μα απαντήσει με μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία. Τι γίνεται με αυτό το θέμα δεν είχατε εσείς την εντύπωση ή την αίσθηση ότι αυτό το τόσο θετικό ίδρυμα και μέσο υπολειτουργεί, εν πάση περιπτώσει δεν το αξιοποιούμε. Ε, έχει μια πολύ περιορισμένη τοπική ίσως οπτική γωνία και δεν έχει ανοίξει τα φτερά του μέχρι αυτές τις χώρες όσο θα έπρεπε. Και ένα άλλο που θα ήθελα να σας πω. Αυτή η διαδικασία κατανοώ ότι θα πρέπει να είναι μια διαδικασία νομιμοποίησης στις χώρες αυτές και θα χρειαζόταν μια στρατηγική ακριβώς ε, που θα αναζητούσαμε συνέργειες και με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιος το ανέφερε αυτό, νομίζω θα πρέπει να διευρυνθεί και θα πρέπει να γίνει κατανοητό που δεν είναι αυτή τη στιγμή ως κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το σταθμίσουμε, ότι δεν είμαστε νησί στην παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δεσμούς και συνεργασία με μια σειρά τρόπων ε, επικοινωνία, εμπόριο. Δεν είμαστε αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Και μάλιστα δεν είμαστε νησί ευημερία και ευκαιριών για το μέλλον. Εάν μας περιβάλλει ένας ωκεανός φτώχειας, μιζέριας και άγνοιας. Λοιπόν, ακριβώς η σχέση της νότιας όχθης με τη βόρεια όχθη της Μεσογείου αποτελεί μεγάλη απειλή για μια μελλοντική Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη να σεμνύνεται ότι είναι αυτάρκης και ε, γύρω-γύρω τι θα γίνουν. Έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένη η σημασία ήδη της Ευρώπης στα διεθνή τεκτενόμενα. Μήπως χρειάζεται νέα αναθεώρηση μετά εκείνη του 2008, γιατί από τότε ξέρετε πόσο νερό έχει κυλήσει κάτω από τις γέφυρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέρος του κόσμου που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και εργάζεται εκεί. Επίσης, έχω την εντύπωση, παρόλο που δεν τα γνωρίζω σε βάθος αυτά, ότι τα προβλήματα της αξιολόγησης των οργανισμών μας θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Νομίζω αναβαθμίζεται ήδη, γιατί αυτοί οι οργανισμοί, οι agencies της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τη χάνουν τη συνένεση εκείνη που θα έπρεπε. Και ορισμένοι που θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι απλώς μια κοινή αγορά, δεν καταλαβαίνουν γιατί έχουμε τόσους οργανισμούς και τόσες προτάσεις. Δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο κοντόφθαλμοι και τόσο μείωπες, γιατί αυτοί που θεωρούν αυτό την Ένωση ένα απλό σύνολο ε, που συνεργάζεται εμπορικά δεν καταλαβαίνουν γιατί έχουμε τόσους οργανισμούς και τόσες δραστηριότητες. Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί και αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και να το ζητούν οι ίδιοι οργανισμοί. Γιατί είναι δύσκολη και κυρία χαλεπή. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε. Α, δεν ξέρω αν θέλουν και άλλοι συνάδελφοι το λόγο. Όχι. Σας παρακαλώ λοιπόν να απαντήσετε και ήδη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας ε, δώσω κάποιες απαντήσεις. Περίπλοκες είναι βέβαια οι ερωτήσεις. Καταρχήν, Ίσως ε, να τοποθετήσουμε εκ νέου στην πραγματική του διάσταση αυτό το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα. Έχουμε, έχει 80 εμπειρογνώμονες που πρέπει να εργάζονται σε καμιά τριανταριά χώρες και η ισχύ των παρεμβάσεών μας είναι σχετικά μικρή. Δεν λέω ότι πρέπει να το εναυξήσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά τις δυνατότητες παρέμβασης για το σύνολο των χωρών αυτών. τα ίδια θέματα που αναφέρατε για το θέμα της ε, πρόληψης, ε, πώς δηλαδή θα μπορούσαμε να προετοιμάσουμε τους νέους ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν όλα αυτά, δηλαδή πιο δουλειά να τους προετοιμάσουμε, τι θα κάνουν αργότερα. Αλλά εδώ έχουμε εταιρικότητα, εταιρική σχέση και το συνεργασία με τις χώρες της νότιας ε, όχθης της Μεσογείου και τις ε, χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Ε, συμπληρωματικότητα μόνο και μόνο μετακινώντας, μετα... τις επιχειρήσεις. Τι είδους εταιρική σχέση θέλουμε να έχουμε και προφανώς αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στην απασχόληση. Τώρα όσον αφορά την απασχόληση σε αυτές τις χώρες, να πω ότι για το 2025 θα πρέπει να δημιουργηθούν 60 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης για να εγγυηθούμε την κοινωνική συνοχή στην νότια όχθη της Μεσογείου. 60 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, εδώ λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των νέων κάτω των 25 ετών στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Τινησία, στην Αίγυπτο, Ξέρουμε ότι σε 10 χρόνια 60 με 80% των θέσεων απασχόλησης θα είναι ίδιες όπως και σήμερα. Το περιεχόμενό τους θα είναι το ίδιο, ε, θα έχει αλλάξει, αλλά πάντα θα έχουμε καθηγητές, νοσοκόμες, ε, ξυλουργούς, ε, εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, ξενοδοχειακούς υπαλλήλους κτλ. κτλ. Το ίδιο ισχύει για την νότια όχθη της Μεσογείου όπως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει όμως να υπάρχουν και ε, νέα προσόντα. Νέα προσόντα σε σχέση με την τεχνολογία, τις επικοινωνίες κτλ. κτλ. Ε, όλα αυτά εξαρτώνται και από τον τρόπο συνεργασίας, τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η δουλειά. Τώρα αυτές τα προσόντα αποκτούνται με περισσότερη μελέτη, πιο μακρές σπουδές. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος. Και το παράδειγμα της Τινησίας μας το δείχνει δυστυχώς με νέους ε, που έχουν το ΜΠΑΚ ε, συν 6 συν 8 ε, χωρίς δουλειά και που δεν φαίνεται να προοδεύσουν ακόμα και αν προχωρήσουν σε περαιτέρω σπουδές προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι ακόμα και αν μιλάμε για την αγορά εργασίας υπάρχουν διάφορες αγορές εργασίας. Ε, η αγορά, η εργασίας των ξυλουργών, των οικοδόμων δεν είναι η ίδια με τους, ε, την αγορά για τους γιατρούς ή για τους νοσοκόμους. Και για διάφορες θέσεις απασχόλησης και δραστηριότητες, σε μια περιφερειακή μάλλον ε, προσέγγιση είναι πολύ σημαντική. Και αυτό γιατί, για να συνδεθεί η ανάπτυξη μιας οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργεί θέση απασχόληση και της κατάρτισης που γίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή το όνειρο του νεαρού την ίση που έχει πτυχίο στη ανώτατη της εκπαίδευση είναι να γίνει δημόσιος υπάλληλο Και μπορούμε πολύ καλά να το κατανοήσουμε αυτό. Πώς όμως θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της δραστηριότητας στην χώρα του και ιδιαίτερα στα βάθη της Τινησίας, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ε, οι νεότερε γενναίε, όπως σας είπα, είναι ιδιαίτερα πολυάριθμε εκεί σε αυτές τις χώρε και θα πρέπει γι' αυτό ίσως να ξανασκεφτούμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν θα πρέπει να μείνει ένα σύστημα ταυτόσιμο με αυτό που υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Τώρα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ κατάρτισης και απασχόλησης, εδώ νομίζω πως ε, θα πρέπει να ε, ενταχθεί και η κατάρτιση διαβίου. Ε, δεν είναι μόνο η αρχική κατάρτιση που θα επιτρέψει για 40 χρόνια ενεργούς εργασιακού βίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ένας εργαζόμενος. Τώρα, όσον αφορά την, την νομιμότητα αυτού του Ιδρύματος, νομίζω πως είναι πραγματική, αναγνωρίζεται εξάλλου από την Διεθνή Τράπεζα, από τις υπηρεσίες, του οργανισμούς ανάπτυξης των διαφόρων κατώμελων και συχνά σε κάθε χώρα μάλιστα αυτές οι διάφορες παρεμβάσεις δεν είναι εύκολο να τι συντονίσουμε. Πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε κάθε φορά την ε, θέση μας. Και απαντώντας συγκεκριμένα στο ερώτημά σα να πω ότι η εντολή του Ιδρύματος, όπως ορίζεται από τον κανονισμό, είναι σωστή και ε, λειτουργεί. Αυτό που μπορεί να λείπει είναι, και επιτρέψτε μου να το πω, είναι η χρηματοδότηση. που δίνει η Ένωση, όχι στο Ίδρυμα, αλλά στις χώρες εταίρους. Αν δούμε τις χώρες του Μαγκρέμπ, στην ουσία ανακυκλώθηκαν οι πιστώσεις που ήδη είχαν προβλεφθεί πριν από το Αραβική Άνοιξη. Δεν υπήρξε καμία σημαντική αύξηση όσον αφορά την ε, κοινοτική αρρωγή προς τις χώρες αυτές. Yes, I would, I would like to start... κύριος θα ήθελα να πω καταρχάς ότι Υπάρχουν πολλές επικρίσεις διερχόνων οργανισμών που παρέχουν τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες και υπανάπτυκτες χώρες. Βρήθη η διεθνής βιβλιογραφία τέτοιων επικρίσεων. Ότι προσπαθούμε να ε, μεταμοσχεύσουμε περίπλοκες τακτικές και τεχνικές για να αλλάξουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα, ιδιαίτερα την επαγγελματική κατάρτιση στις χώρες αυτές. Γιατί το λέω αυτό. Θέλω να πω στη συνέχεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επί σειρά ετών έχει αναπτύξει δύο πολύ αποτελεσματικά μέσα και εργαλεία και όχι τόσο περίπλοκα και τα εφαρμόζει που είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, δεξιοτήτων βέβαια που όταν εφαρμοστεί στην εκάστοτε χώρα υιοθετείται και γίνεται εθνικό πλέον πλαίσιο και το δεύτερο είναι ο θεσμός των κοινωνικών εταίρων Αυτά τα δύο λοιπόν είναι οι δύο πρώτες στρατηγικές και μέσα που προσπαθεί το Ίδρυμά μας να εφαρμόσει στις περισσότερες ε, δικαιούχες ε, χώρες. Και αυτό ισχύει και για τις χώρες Βορειοαφρικής. Οπότε, το ερώτημα για την τεράστια αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων και μάλιστα υψηλού επίπεδου μπορεί να ισχύει μέρη στις χώρες αυτές, όπως είπε και ο συνάδελφος. Υπάρχουν ε, ειδικέ δεξιότητες που μπορεί να χρειάζονται, ε, ε, αλλά θα πρέπει να συνεργάζονται οι κυβερνήσεις, ε, οι ε, εργοδότες, εκείνοι που εκπαιδεύουν και παρέχουν αυτή την ε, υπηρεσία, θα πρέπει να είναι αρκετά ρεαλιστική η προσπάθεια για να αποδίδει και να αναπτύσσεται το ανθρώπινο δυναμικό με τρόπο αποτελεσματικό. Ένα άλλο θέμα που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο εδώ είναι η δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να ε, προωθήσει τη δημιουργία ενδογενών ικανοτήτων ε, για να ασκούν και να χαράσουν πολιτικές οι ίδιοι. Ε, γιατί ρωτήσατε για τις μεταρρυθμίσεις. Πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης που να ταιριάζουν με τις ανάγκες τους, να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης ε, που να συνάδουν με προγράμματα σπουδών ε, εκπαιδευτικά. Αφού λοιπόν επένεσα τόσο πολύ το θεσμό των κοινωνικών εταίρων, θα ήθελα να πω στα μέλη της Επιτροπής σας ποια είναι η πραγματικότητα στις αναπτυσσόμενες και επανάπτυκτες χώρες ως προς τους κοινωνικούς εταίρους σε στρατηγικές συνεδριάσεις τι συμβαίνει συνήθως. Οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων κυριαρχούν σε όλη τη συζήτηση. Καπελώνουν πολλοί. Οι εργοδότες δεν λένε και πολλά και αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Μια κρίσιμη λοιπόν δράση σε αυτή την περίπτωση που έχει εφαρμοστεί σε κάποιε υπανάπτυκε χώρες είναι να εκπαιδεύει τους εργοδότες να συμμετέχουν σε αυτές τις σκέψεις με τρόπο αποτελεσματικό και να αρθρώνουν ε, τις ανάγκες τους, να τις παρουσιάζουν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά και να λέγουν τι τους χρειάζεται για να έχει σημασία και νόημα και αποτέλεσμα η κοινωνική εταιρική σχέση αυτή ο κοινωνικό διάλογο. Γι' αυτό θα πρέπει να λέγουν εκείνοι που έχουν τις ανάγκες, τι ανάγκες έχουν για να ακολουθεί και η εκπαίδευση και να κουμπώνει με την αγορά εργασίας. Σε σχέση με τη δεύτερη παρέμβαση του κυρίου Σέρκας, η απάντησή μου περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα της έκθεσής μου, σας παραπέμπω και δίνω μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση του Ιδρύματός μας όχι τόσο πολύ από την πλευρά της λογοδοσίας, αυτό κατά την άποψή μου είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον ως λειτουργία μιας αξιολόγησης είναι διαγνωστική ικανότητα. Να εντοπίζεις, δηλαδή να επισημαίνεις ε, κάποιες ελλείψεις, ε, δυσλειτουργίες και να μην περιμένουμε να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα, αλλά να ενημερώνουμε με ένα feedback, μια παρακολούθηση συνεχώς. Δεν περιμένουμε να ολοκληρωθεί ένα έργο για να διαπιστώσουμε ή να συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι πήγε στραβά. Bien, il nous reste euh, à vous remercier. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν. Κύριε Ντεμεζιέρ, ε, σίγουρα θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να σας δούμε εδώ ή στο Τωρίνο. Και κύριε Παλαιοκραστά, θα σας ευχαριστήσουμε για τον απολογισμό δραστηριοτήτων. Εγώ πήγα αυτοπροσωπώ στο Τωρίνο και πραγματικά συνειδητοποιώ πόσο πολύτιμο είναι το Ίδρυμα Κατάρτισης γιατί συμβάλλει στην όλη δυναμική της ε, ηγεσία το Έτσι, ε, η επιτυχία την είναι συνάρτηση και της ποιότητας της δουλειάς όλων των συνεργατών σας. Είναι καθοριστικός ο ρόλος σας, τόσο από τι βέλτιστε δυνατέ προποθέσει να λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα στο πλαίσιο όλων των συζητήσεων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντω, ε, το όλο θέμα τη σχέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με του Οργανισμού, το θέμα του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τους οργανισμούς, όλα αυτά τα στήματα δείχνουν ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και η πραγματογνωμοσύνη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αίρισμα για τις ε, πρωτοβουλίες που υλοποιούνται επί τόπου στις χώρες. Για το, ως προς τη νέα σας εντολή θα έλεγα το εξής. Όταν κάποιος οργανισμός ε, κατόπιν αιτήματος επιτροπής μας ή κάποιας άλλης ε, δημοσιεύει μία έκθεση, ε, σίγουρα πρέπει να χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει τις νομοτεχνικές εργασίες μας και νομίζω ότι ο εμπειρογνώμονα που θα έχει συντάξει αυτή την έκθεση, καλό θα ήταν να έρχεται εδώ επί τόπου στι συνεδριάσει μα για να μα παρουσιάζει την έκθεση του. Αυτό θα συνιστούσε θεμενή αξία. Σα ευχαριστούμε πάντω για την ενημέρωση και στο επανειδήν. Ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο. Δεν θα διακόψουμε για πάρα πολλή ώρα τις εργασίες μας. Μην φύγετε παρακαλώ από την αίθουσα. Όλοι οι δικοί μας εδώ στο Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι καθοδόν και θα φτάσουν σε λίγα λεπτά όπου και θα εξετάσουμε την έκθεση της κυρίας Χάρκη. Μην αποχωρήσετε σας παρακαλώ πολύ. Ε, ήρθατε ακριβώς την ώρα που έπρεπε κυρία Χάρκιν, καλώς ορίσατε και πάλι. Παρόλα αυτά θα περιμένετε κι εσείς, ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι πιο σωστό για τις υπόλοιπες ε, πολιτικές ομάδες ε, και το τους συνεργάτες σας από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες για να έρθουν. Ο κύριος Νταγντά έρχεται, κυρία Χάρκιν ήρθε. Θα περιμένουμε λίγα λεπτάκια για να έρθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Παρακαλώ. Bon, écoutez, euh, on va commencer, je euh, Αρχίσουμε, νομίζω. Και αρχίζοντα θα προσελκύσουμε και την κυρία Κορνέλισεν. Ότι δεν γίνεται να περιμένουμε και σάι. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων για την ε, κυρία Κορνέλισεν λυπάμαι, αλλά θα ακούσουμε την κυρία Χάρκιν. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, για την έκθεσή σας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την περίοδο 2014 έως 2020. Πριν σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ε, ότι θα συζητήσουμε με την Επιτροπή Άγκρη για το θέμα αυτό. Συζητήσαμε, συγγνώμη, με την Επιτροπή Άγκρη. Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι φαίνονταν στην αρχή και άρα προς το παρόν δεν γνωρίζουμε την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις δύο συναρμόδιες επιτροπές πάντως γνωρίζουμε το περιεχόμενο του σημειώματος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ε, σας ακούμε κυρία Χάρκη. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, μετά τις συζητήσεις με την Επιτροπή Αγρί. Ήθελα μόνο να τα υπενθυμίσω για τους συναδέλφους να ενημερωθούν για τις ε, τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε ε, συσκεφθεί διάφορες φορές με τον εισηγητή, τον κύριο Άλβαρες, για να καταλήξουμε σε κάποιο είδους συμφωνία. Δεν κατέστη αυτό δυνατό. Στην συνεδρία των συντονιστών της Επιτροπής Απασχόλησης αποφασίσαμε ότι η Επιτροπή μας θα επιδιώξει πλήρη αρμοδιότητα για το θέμα αυτό και δεν είμαστε υπέρ χορήγηση αποκλειστικής αρμοδιότητας στην Επιτροπή Γεωργίας ε, για τα σχετικά με αυτή την αρμοδιότητα τα υποζητήματα της έκθεσης. Σανθήκαμε με τους κυρίους Αντόρ και Τσόλος. Ε, ήταν και οι πρόεδροι των δύο συναρμοδίων επιτροπών, οι συγητές, σκιώδης και τα λοιπά, για να δούμε αν τελικά ε, θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν κατέστη δυνατό. Κάναμε μια ενδελεχέστατη συζήτηση για όλα τα ζητήματα, αλλά δεν κατέστη δυνατό να καταλήξουμε σε συμφωνία. Κατόπιν είχε προβλεφθεί σύσκεψη για τους συντονιστές για την Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, τελικά μετατέθηκε για την Πέμπτη και τώρα πάλι ακυρώθηκε. Η σύσκεψη των συντονιστών δεν ξέρω αν έχετε άλλη ενημέρωση, Πρόεδρε, αλλά εγώ αυτά ξέρω. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση και μάλλον το θέμα θα πάει στη διάσκεψη των ε, Προέδρων για να ληφθεί μια απόφαση. Οι σκιώδεις ε, μετά από τη σημερινή συνεδρίαση θα συσκεφθούν ε, για να δούμε αν υπάρχουν νέες προτάσεις και για να αποτελματωθεί η συζήτηση. Μέχρι στιγμή σα είπα πόσο δύσκολο ήταν αυτό, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Μπορώ να σα πω πάντω ότι η Επιτροπή μα ανέθεσε ένα εξαιρετικά δυσχερέ έργο. Ε, είμαι μέλο ε, και στην Άγκρη, πληρωματικό μέλο τη Επιτροπή Γεωργία και μπορώ να σα πω ότι ε, ούτε στην Άγκρη θέλουν αυτή την έκθεση γιατί θεωρούν ότι είναι ο δούριο ύπο. και η μάρκα ΣΕΡ Αναγκάστε να τη δεχτεί για άλλους λόγους, για λόγω άλλων εκθέσεων. Η Άγκρη εν ολίγησε θέλει να διατηρήσει ε, την ε, αρμοδιότητά της, αλλά είναι δίλητη το δώρο και το ξαναλέω. Λοιπόν, αναφέρει η Επιτροπή τη δυνατότητα τη, να αποδοθεί στην άκρη το 83% του ταμείου. Αυτό φυσικά ε, συνιστά πρόβλημα. Τέλος, η Επιτροπή ε, Περιφερειών στη δική του νομοθέτηση αναφέρουν ε, λυπούμεθα για την ε, απόφαση βάση τις οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς ε, οι γεωργοί. Δεν υπήρξε υποστήριξη να συμπεριληφθούν ε, οι γεωργοί μέσα στην έκθεση κατόπιν πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα ε, περί αρμοδιοτήτων ε, όμω αυτό παρεμποδίζει την όλη διαδικασία διότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μέχρι ότου ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα. Α κάνω παρόλα αυτά κάποια σχόλια γιατί θέλω να ακούσω και την άποψη των συναδέλφων. Εγώ είμαι πραγματικά υπέρ ε, του να καλυφθούν ε, και οι αυτοαπασχολούμενοι και όσοι ε, έχουν προσωρινές θέσεις εργασίας μέσω των γραφείων ευρέσεω εργασία ε, και να καλυφθούν και οι γεωργοί, αλλά όπως ε, επί τη ίδια, της ίδιας βάσης, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, δηλαδή ε, η παγκοσμιοποίηση, οι αλλαγέ αλλαγές που διαφέρουν ανακλάδο, αν συγκρίνουμε τη γεωργία με την αυτοκίνητο βιομηχανία κτλ. Έχω πλήρη επίγνωση της ιδιαίτερότητα του κλάδου, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορέσει αλλιώ να λειτουργήσει το Ταμείο σωστά στην πράξη και θα πρότεινα το εξή. Εάν καταλήξουμε τελικά σε συμφωνία και τεθεί το ζήτημα των γεωργών, σε περίπτωση απώλειας ε, με τις απασχόλησης. Ε, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα μπορούσε να καλύψει τις οικογένειές τους. Αυτό υπάρχει ήδη μέσα στην έκθεση αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το ταμείο θα πρέπει να είναι το βασικό εργαλείο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και, είμαι, και ξέρω εκ των έσω ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για αυτό το θέμα στην Επιτροπή Άγκρη σε σχέση τώρα με την άλλη πρόταση Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά ε, με τα κριτήρια της απροσδόκητης κρίσης ε, τα οποία διαφέρουν από τα κριτήρια που διεύουν την τωρινή κρίση που δεν είχαν ε, επεκταθεί από το Συμβούλιο και θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο για να σα εξηγήσω ότι έχει κατά Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή σκέφτονται το εξή αν έχουμε μια, ε, ένα θέμα όπως αυτό του ηφαιστείου και της ε, στάχτης ε, και έπρεπε, χρειάστηκε να κλείσει μια αεροπορική εταιρεία λόγω των προβλημάτων και των ζημιών ή τέλος πάντων να υπάρχουν απροσδόκητες πλημμύρες όπου σε κάποιες χώρες έκλεισαν εργοστάσια, τέτοιου είδους απροσδόκητες κρίσεις που δίνουν, που επισύρουν απώλεια πολυάριθμων θέσεων απασχόλησης με αυτόν τον απρόβλεπτο τρόπο. Τέλος πάντων προτείνεται να συμπεριληφθεί και αυτό και να έχουμε μια νέα δέσμη κριτηρίων μέσα στην έκθεση. Ε, αλλά Εκεί αλλάζει και η πρικοδότηση του Ταμείου. Δεν έχουμε πλέον τους ίδιους κανόνες τα 500 εκατομμύρια που πρέπει να εκταμιευθούν μέσα σε τέσσερι μήνες κτλ. κτλ. Όμως, ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε ε, επίγνωση του ότι δεν έκαναν χρήση τα κράτη-μέλη στο μέτρο ή με τη συχνότητα που προβλέπαμε στην αρχή. Το χρονικό λοιπόν ζήτημα επανέρχεται. Ο μηχανισμό που έχουμε στην ε, διάθεσή μας κατά τη γνώμη μου δεν μας επιτρέπει να τροποποιήσουμε πολύ περισσότερο το χρονοδιάγραμμα, οπότε Ποιε είναι οι λύσει, ε, οι εναλλακτικέ. Πρώτον, να ε, πιέσουμε τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε με το που υποβάλλουν αίτηση για ενεργοποίηση του Ταμείου να αρχίζουν και τη διαδικασία και να εφαρμόζουν τα μέτρα. Κάποιοι, κάποιοι θα αντιτάξουν ότι δεν έχουν κονδύλια για να εφαρμόσουν τα μέτρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βοηθάει τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να υπομισθούν τι ευθύνε και να βοηθήσουν του εργαζομένου του. Και κάτι άλλο που ανέφεραν ένα-δύο συνάδελφοι και ξέρω το έχω ξαναπεί, αλλά το ξαναλέω διότι ε, μπορεί να έχουν προκύψει νέες ιδέες, ε, να υπάρχει ε, ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού δηλαδή για το Ταμείο. Εν τη αυτή περιπτώσει θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για την εφαρμογή των μέτρων. Αυτά έχουν γίνει μέχρι στιγμή και δεν θα επεκτάθω, Πρόεδρε. Θα ακούσω μόνο του συναδέλφου. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ και μετά οι Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να αρχίσω με μια ερώτηση που παραμένει αναπάντητη. Ως προς την επιστολή σας ε, προς το Συμβούλιο. Για μένα η απάντηση που δόθηκε ήταν κάτι που μου προξένησε έκπληξη. Γιατί λέει το Συμβούλιο ότι αυτό το καιρό γίνεται μια συζήτηση που θα πρέπει να λάβει υπόψη τη την κρίση για το Ταμείο αυτό. Αλλά αν γινόταν ε, με τέτοιο τρόπο ε, θα διακύβευε, μάλλον θα υποθήκευε τη μελλοντική συζήτηση για το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Τι θα πει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Μήπως εσείς ξέρετε τίποτα περισσότερο ε, πώς να ερμηνευτεί ε, αυτή η απάντηση και τι επιπτώσεις έχει για το δικό μας μέλλον και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το θέμα συμπερίληψης των γεωργικών θεμάτων έχει λήξει ή αν παραμένει ακόμα ανοιχτό. Έχει κανένα νόημα να το συζητούμε. Δεν είναι καλή απόφαση πιστεύω. Να καλύψουμε από το ταμείο αυτό και τη γεωργία. Διότι, κατά την άποψή μου, στην κοινή αγροτική πολιτική έχουμε πολλά μέσα και και θα ήταν ίσως σκοπιμότερο να στραφεί εκεί η γεωργική πολιτική και να μην αναμειχθεί με το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ένα τρίτο που ήθελα να αναφέρω είναι η προσωρινή ενίσχυση από το Ταμείο. Φαίνεται αυτή η διετία είναι πολύ μακρύ χρονικό διάστημα ε, για να απαντήσουμε σε μια κατάσταση κρίσης. Είτε για την παγκοσμιοποίηση, είτε για την κρίση αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή, ε, πρέπει να βρούμε μια απάντηση για αυτό το θέμα. Και συμφωνώ απολύτως ότι το βασικό θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τη γεωργία σε αυτό το, θέ, το ταμείο που δεν έχει θέση εκεί. Ο κύριος Νταρντέν και μετά ο κύριος Τόμας Μαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κάποιες ε, σκέψεις που τις έχω ήδη εκφράσει σε παλιότερες ε, συναντήσεις, αλλά είναι ευκαιρία για να επανέλθουμε. Καταρχήν, νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε την ε, λύπη μας, γιατί ότι δεν καταφέρνουμε να κατανέμουμε τις αρμοδιότητες και να διευκρινίσουμε αυτά τα προβλήματα. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται, δεν το έχουμε καταφέρει αυτό και μάλιστα θα έλεγα ακόμα και ότι μας εμποδίζει αυτό να θίξουμε την ουσία. Είναι πραγματικά σημαντικό να θίξουμε την ουσία, γιατί δεν είναι δεδομένα όλα αυτά. Καταρχήν να μιλήσουμε για το θέμα των γεωργών. Είχα την ευκαιρία να εκφραστώ εξ ονόματος της ομάδας μας και πιστεύω πως είναι κακό να υπάρχει ένα ταμείο δύο ταχυτήτων με δύο ε, δυνατότητες ε, που περιορίζει τις δυνατότητες και τις διαθεσιμότητες για το σύνολο των εργαζομένων. Γιατί τα κονδύλια που θα, θα περιορίζονταν από ένα ανώτατο όριο ήταν ε, τεράστια σε σχέση με το σύνολο του ταμείου και αυτό μου προκαλεί ανησυχίες. Και πιστεύω επίσης ότι σε σχέση με το συγκεκριμένο με εργαλείο θα ήταν πολύ πιο απλό το πράγμα και πιο διαφανές όσον αφορά τα συγκεκριμένα κονδύλια στον προπολογισμό. Σε μεγάλο βαθμό ε, συμφωνεί με τα όσα έχω ήδη πει εδώ ή στο πλαίσιο των δημοσιονομικών εργασιών να διευκρινίσει, μπορούσε να διευκρινίσει τα πράγματα και να αυξήσει τις δυνατότητες εκτέλεσης, ανταπόκρισης στα αιτήματα και αναμφίβολα είναι ένα από τα δύνατα σημεία αυτή τη στιγμή του κονδυλίου. Και εν πάση περιπτώσει είναι κάποια από τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί. Οι επικρίσεις κάποιες φορές είναι υπερβολικές, αλλά είναι σαφές ότι η πτυχή του καθυστέρησης πούμε, των απαντήσεων είναι ε, σημαντική. Ε, και, επίσης η ταχύτητα εκτέλεσης είναι ε, αργή. Και μόνο ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις επικρίσεις και αυτές τις αδυναμίες ε, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το, το ταμείο αυτό, το οποίο έχει χρησιμότητα. Επ' αυτό δεν έχω αμφιβολία. Πολλές φορές παρεμβαίνοντας από διάφορες χώρε εξηγούσαν πώς το χρησιμοποιούν στις χώρες τους και μετά ήμουν ακόμα πιο πεπισμένος για την χρησιμότητα και για τη σημασία των εργαζεμένων που έπεσαν θύματα αναδιαρθρώσεων συχνά λόγω κρίσης. Όταν θέλουμε να καταργήσουμε και όταν θέλουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το κριτήριο κρίσης, εγώ πιστεύω πως είναι ένας βασικός δείκτης της ελαφρότητας, για να μην πω τίποτα παραπάνω, ορισμών κρατών σε σχέση με την ε, βούλησή τους για διατήρηση του Ταμείου. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να αφήξουμε αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να προτάξουμε όλα τα σωστά επιχειρήματα έτσι ώστε να ενισχυθεί και να ευνοηθεί η διατήρηση αυτού του, του Ταμείου. Ο κύριο Τόμας Μάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ακριβώς να επενέσω την κυρία Χάρκιν ε, και να συμφωνήσω και το έχουμε πει στους συντονιστές επανειλημμένα και στους κοιόδης ηγητές. Δεν μπορεί τώρα να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία ή να την εκμεταλλευτεί η Επιτροπή Γεωργίας για να μπει σε αυτό το μικρό ταμείο. Και εγώ έχω αγρότες στην εκλογική μου περιφέρεια. Κανείς δεν μου ζήτησε επιπλέον λεφτά από αυτό το ταμείο. Έχουμε τόσα ταμεία στα γεωργικά. Αν δεν γίνεται, να το φροντίσουμε αλλού στη νέα χρηματοδότηση της γεωργίας μπορεί να γίνει αυτό κάλλιστα αν το θέλουμε. Θυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε από τον κύριο Παρόσο και στην αρχή είχαν αντισταθεί με νύχια και με δόντια τα κράτη-μέλη και πολλοί είχαν λάβει τι αποστάσει του. Ναι, Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, ωραίο το μήνυμα, αλλά τι θα βγει από αυτό. Και μήπω είναι χρήματα που θα βγουν από το Κοινωνικό Ταμείο και πάλι. μήπω είναι μια φούσκα μήπως είναι αντικατοπτρισμός. Τελικά η πραγματικότητα έδειξε ότι λειτουργήσε σωστά στην πράξη και χαρήκαμε γι' αυτό. Να βοηθήσουμε εταιρείε που έχουν μεγάλα προβλήματα αναπροσαρμογής και τους είπαμε ότι δεν τους αφήνουμε στη μοίρα τους. Να έχουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα και σημαντικό για να απαντήσουμε στην παγκοσμιοποίηση. Και πολλά λειτουργήσαν σωστά τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι κυρία Ματέρα που στο, στην Ολομέλεια κάθεται δύο θέσεις πιο ε, πέρα από μένα και πάντα το έλεγε αυτό στις μονόληπτες και δίλεπτες ε, τοποθετήσεις στην Ολομέλεια. Για ποιες χώρες πρόκειται. Το θέμα δεν είναι ότι έχουμε λεφτά και τα μοιράζουμε κατά το δοκούν. Όχι. Οι άνθρωποι δικαιούνται να τους στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης και είναι σωστό αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξή, Μάριαν. Στα κράτη-μέλη τι γίνεται. Συμφωνούν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουμε το ταμείο αυτό, να το εφαρμόσουμε. Αν υπάρχουν επιφυλάξεις, πώς εκφράζονται, με ποιο τρόπο και ποιες δυνατότητες υπάρχουν. Γιατί δεν συμφωνούν απολύτω οι πάντες με το Συμβούλιο. Ποια είναι τα κράτη-μέλη που διατηρούν μεγάλες επιφυλάξεις και γιατί. Και μπορούμε να τα μεταπίσουμε διότι χρειάζονται περισσότερα η βοήθεια οι άνθρωποι από μια μικρή ε, αλληλεγγύη ή με καλά λόγια ή αν κάνουμε πορείες διαμαρτυρίας. Θα πρέπει και συγκεκριμένα να τους δίνουμε στην πράξη το μήνυμα ότι έχουν μέλλον. Ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε τα κριτήρια, αλλά όχι να το απορρίπτουμε σε αυτό το ταμείο. Ευχαριστώ. Πριν ε, δώσω την προεδρία στην κυρία Σρότερ, γιατί πρέπει να φύγω. Ε, θέλω να πω και εγώ μερικά λόγια στη συζήτηση αυτή. Η έκθεση της κυρίας Χάρκιν εγγράφεται στο πακέτο των δημοσιονομικών προοπτικών και για την Επιτροπή μας είναι εξαιρετική σημασία γιατί βλέπουμε ότι θίγει διάφορα σημεία και είναι ένας από τους μοχλούς πίεσης που έχει η Επιτροπή μας για να μπορέσει να διαβιβάσει αυτά τα μηνύματα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση απαντά στον κοινωνικό αντίκτυπο από την παγκοσμιοποίηση και την αλλαγή του κόσμου που έχουμε βαφτίσει παγκοσμιοποίηση είτε είναι το κριτήριο παγκοσμιοποίηση είτε η κρίση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι συνέπειες που υφίστανται οι πιο ευάλωτοι από τις εξελίξεις αυτές. Εμείς που διαφωνούμε τώρα με την Επιτροπή Γεωργίας ή που συγκρουόμαστε. Και αυτό δεν θα μας εμποθήσει να αντιμετωπίσουμε και τα άλλα θέματα αλλά είναι εύγλωτη για τον τρόπο με τον οποίο προχωρήσαμε στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με διάφορες χώρες εταίρους μας. Χωρίς να ληφθεί υπόψη η ε, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση αυτών των συμφωνιών και ότι δεν είναι δίκαιη η συναλλαγή αυτή και ορθή. Και επειδή θα προχωρήσουμε και σε άλλες τέτοιες συμφωνίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην δεχόμαστε ότι να είναι. Δηλαδή, μέσω αυτής της έκθεσης να βάλουμε κάποια κριτήρια και να έχει θέση το κοινοβούλιο ότι στο μέλλον δεν θα δεχθούμε πλέον υπογραφή τέτοιων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Αυτή τη στιγμή το άρθρο 9 της συνθήκης και επανέρχομαι πάντα σε αυτό, δηλαδή η κοινωνική διάσταση και απασχόληση δεν εφαρμόζεται και με τρόπο πάρα πολύ αυστηρό δεν αξιολογείται. Γιατί αν είναι αυτή η περίπτωση Μάλλον αν είχε ισχύσει κάτι τέτοιο δεν θα είχαμε υπογράψει με τη Μερκοσούρα αυτά που υπογράψαμε. Για τους δε αγρότες αυτό που φαντάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τελείως απαράδεκτος λύση. Απαράδεκτο. Βλέπουμε ποια είναι η φτώχεια, η ανεργία στην Ένωση και στα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή λέει κάποια κράτη ε, μέλη δεν θέλουν να εκτεθούν σε σχέση με το προϋπολογισμό της Ένωσης για τη Γεωργία, που ξέρουμε ότι θα περιοριστούν τα χρήματα πλέον, έρχονται πλαγίους και βάζουν χέρι στην τσέπη του κοινωνικού ταμείου ή του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εκεί είναι μια δεύτερη διάσταση που για μένα τελείω τελείως σημαντική, ουσιώδης. Λυπάμαι που παρά τις τόσο καλές επαφές που είχαμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε με τους συντονιστές. Η δαμόκλια σπάθη της μεγάλης διάσκεψης των προέδρων που θα κληθεί λέει να αποφανθεί και καλό είναι να το λύνουμε μεταξύ μας πριν φτάσει μέχρι εκεί. Και ένα τελευταίο που θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη μας στην έκθεση Χάρκιν είναι οι επικρίσεις για το Ταμείο, το ίδιο. Αναφερθήκατε κι εσείς σε μερικές. Είναι γεγονός αυτό, είναι τελείως ανυπόφορο πια. Στο Συμβούλιο δεν κατάφερε να απεμπλακεί η ε, παράταση ε, του μηχανισμού για την κρίση. Που ακόμα και η Δανία ε, το αξιοποίησε για τη χώρα της. Και βλέπουμε ότι η κοινωνική κατάσταση που συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση ή την κρίση μέρα με τη μέρα επηρεάζει εκατοντάδες ε, μισθωτούς της χώρες μας. Δηλαδή, αυτό το θέμα πρέπει να το δούμε. Χρειαζόμαστε μένα αυτό το ταμείο, αλλά που να λειτουργεί. Γιατί έτσι όπως έχει σήμερα δεν λειτουργεί καλά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξανανοίξει η μάχη για το ειδικό κονδύλι του προπολογισμού για να επιταχυνθεί αυτό το να αλλάξουμε τις προθεσμίες στο Κοινοβούλιο δεν θα επιταχύνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και θέμα της θέσης του προπολογισμού. Άλλο θέμα τώρα. Αυτοί, ε, αυτά Είναι πολύ καλή η πρόταση, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται και ε, από μια σκέψη για τα κατόφια. Δηλαδή, αν πρέπει να βρούμε 500 αυταπασχολούμενους στην ίδια περιφέρεια για να είναι δικαιούχοι, παράδειγμα, μια περιφέρεια που πλήττεται από ε, τις αλλαγές στη βιομηχανία δέρματος. Πού να βρεις 500 βυρσοδέψες στην ίδια περιοχή αυτοπασχολούμενους για να τους ενισχύσεις. Αυτό είναι ζήτημα. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι πέρα από τους αυτοαπασχολούμενους η δυνατότητα που θα μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρουσα να ενταχθούν στους δικαιούχους από το Ταμείο αυτό ε, κάποιοι μισθωτοί που οργανώνονται και ε, αναλαμβάνουν την επιχείρησή τους που κλείνει υπό μορφή συνεταιρισμού. Καλό θα ήταν να μπει αυτό στην νομοθεσία και θα ανοίξει το δρόμο για τους ίδιους τους εργαζομένους να το αξιοποιήσουν βεβαίως με την επιφύλαξη ε, να ενισχυθεί χρηματοδότηση. Δηλαδή, αν οργανωθούν οι εργαζόμενοι να αναλάβουν την βιομηχανία τους ή την επιχείρησή τους, δεν θα πρέπει η χρηματοδότηση να έρχεται μετά από δύο χρόνια. Και τελευταία παρατήρηση, το έχω πει επανειλημμένα εδώ στην Επιτροπή, αλλά έχω λόγο να το πω, να δούμε με ποιο τρόπο αυτή η πολιτική ενδεχομένως να αντιφάσκει με την πολιτική ανταγωνισμού. Δηλαδή, Πώς μπορεί αυτή η πολιτική να ε, χρησιμοποιηθεί ως ε, αντιστάθμισμα της μετεγκατάστασης κάποιων πολυεθνικών που δεν έχουμε κανένα λόγο να εθαρρύνουμε. Ιδού επιγραμματικά και με τη μορφή καταλόγου τα όσα είχα να σας πω και θα αποχωρήσω γιατί δυστυχώς πρέπει να φύγω και θα δώσω την προεδρία στην κυρία Σουρέτερ αλλά προηγουμένως Κύριε Σμπέν. Yes, I just want to um, uh, raise uh, another. Εγώ ήθελα να αναφέρω έναν άλλο λόγο για τον οποίο πιστεύω πως αυτό το ταμείο δεν είναι κατάλληλο για τη Γεωργία. Και νομίζω ότι αυτό μάλλον εξηγεί και γιατί και η Επιτροπή Γεωργίας θεωρεί ότι μπορεί να είναι ένα δηλητηριασμένο δώρο. Εγώ μιλάω ω ίδιος, ως αγρότης ο ίδιος. γιατί οι επιδοτήσεις, ε, επιχειρήσεις συγγνώμη, μπορεί όντω να καταρρεύσουν σε μια βραδιά, αλλά δεν καταραίουν επί τη βάση μιας εμπορικής συμφωνίας. Είναι μάλλον ε, ένας πόλεμος ε, ευθορά. Έχει να κάνει περισσότερο ισολογισμός και όχι το τι κερδίζεις χρόνο με το χρόνο. Δέκα χρόνια περίπου παίρνει το να μείνει χωρίς δουλειά ένας Γιώργος και είναι πολύ σχεδόν σίγουρο ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να να φτιάξει έτσι την ε, αίτημά του ώστε να μπορεί να τηρεί όλα τα κριτήρια. Λέτε ότι μπορεί να πάρει ένα σωρό χρήματα, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει να το καταφέρει λόγω αυτής της φθοράς που όπως σας είπα ε, ε, υπάρχει. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα της ε, της ε, εξάπλωσης, μάλλον της διάσπασης της γεωργικής γης σε πολλά μέρη στην ίδια χώρα. Ε, δεν είναι δηλαδή πάντα ένα, μια γεωργική εκμετάλλευση σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Είναι κατακαιρματισμένα τα αγροκτήματα και μπορεί να είναι τόσο δύσκολο, είναι τόσο πολύ κατακαιρματισμένα που είναι δύσκολο να μπουν, να μπουν όλα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καλύτερα είναι να χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά τα κονδύλια της ανάπτυξης υπαίθρου και όχι αυτό εδώ το ταμείο. Και αυτό εδώ το ταμείο να μπει στη μέση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα πω πολλά για τους αγρότες, Θα έχουμε ξανασυζητήσει. Και νομίζω πως είναι σαφές ότι στην Επιτροπή αυτή και μάλλον και σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο υπάρχει πλειοψηφία να μην συμπεριληφθούν εδώ οι, οι γεωργοί. Και πιστεύω ότι η αντίσταση στο Συμβούλιο θα γινόταν ακόμα χειρότερη. Υπάρχει ήδη αρκετή αντίσταση και αυτό με ανησυχεί. Το να συμπεριληφθούν όμως οι γεωργοί εκεί θα μείωνε πολύ περισσότερο τις πιθανότητες. Εμείς ως πράσινοι όσον αφορά ένα νέο ε, ταμείο συνοχής ε, ε, θα ήμασταν υπέρ του να συμπεριληφθεί ένας μηχανισμός ε, ε, ταχείας αντίδραση και αλλά αν δεν υπάρξει εκεί πλειοψηφία θα ήθελα να υποστηρίξω μια συγκεκριμένη γραμμή στον προϋπολογισμό ως εναλλακτική γιατί εμείς οι πράσινοι πιστεύουμε πως δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, κανένα ταμείο εκτός του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και αν κάποια ταμεία δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται και έχουν υποεκτέλεση, τότε θα πρέπει να απορροφηθούν από άλλα ταμεία. Εμεί στο Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται να αποφασίζουμε για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση μεμονωμένα, γιατί όσο και αν είναι ενδιαφέρουσες και συγκεκριμένες οι διάφορες υποθέσεις όσο και αν τα κάλυπτε όλα αυτά ο τύπος θα ήταν καλύτερο για τους γεωργούς η Κομισιόν να αποφασίζει και εμείς να επιβλέπουμε. Τώρα, ανησυχώ για την θέση των κρατών μελών. Α, όντως θα πρέπει το ETF να γίνει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό και μέσα στην τρέλα που επικρατεί για τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές πλαίσιο κάπως μπορεί και αυτό να υλοποιηθεί και υπάρχουν και κάποιε χώρε όπου γίνονται εκλογέ και μπορεί οι κυβερνήσει που θα προκύψουν να συμφωνούν μαζί μα. Κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ήμασταν από αυτού που όταν έγινε η συζήτηση ουσία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο λέγαμε ότι θα ήταν πολύ καλύτερο και σίγουρα θα ήταν μια πιο μακροπρόθεσμη λύση, μακρόπνοη λύση, αν ε, αποφεύγαμε αυτού του είδους ε, τις ε, θεραπείες, όπως αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Πέρα από τα διορθωτικά μέτρα, εμείς προκρίνουμε μεγαλύτερη κοινωνική ασφάλιση, καλύτερη προστασία των εργαζομένων κατά των πολυεθνικών, προστασία των ε, μισθωτών. Ε, επ' αυτού νομίζουμε πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική των κρατών μελών. Τέλος πάντων, ως προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής ε, στην παγκοσμιοποίηση και δοθεί στις βαρύτα της κρίσης που ζούμε όλοι, πιστεύουμε... Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε καλύτερη πρόσβαση για τους ιονί δικαιούχου. κυρίως ε, για τις πιο ευάλωτες ε, χώρες, αυτές δηλαδή που λαμβάνουν ήδη χρηματοοικονομική βοήθεια. Σε ποσοστό 35% προβλέπεται η συγχρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι βασικό κόλλημα για κάποιες χώρες, κυρίως ε, στις χώρες όπου αυξάνεται ραγδαία το ποσοστό των ανέργων. Γι' αυτό προτείνουμε και θα επαναλάβουμε την πρότασή μας ε, το ποσοστό συγχρηματοδότησης ο πλευρά κρατών μελών να μειωθεί και να παραμείνει στα τωρινά επίπεδα. Σχετικά με την συμπερίληψη ή όχι των γεωργών, πιστεύουμε, όπως ακούσαμε και από συναδέλφους, ότι θα έπρεπε Ε, αυτοί που υπέγραφαν τις διμερεί εμπορικέ συμφωνίε θα είχαν προβλέψει τι αρνητικέ κοινωνικέ επιπτώσει και όχι να τι διορθώνουμε τώρα μέσα από αυτό το ταμείο. Να προλαβαίνουμε και όχι να διορθώνουμε δηλαδή. Eh, e, τώρα οι γεωργοί λοιπόν δεν πρέπει να καλυφθούν από το ταμείο, κατά τη γνώμη μας. μεταξύ άλλων επειδή υπάρχουν ήδη άλλα μέσα και ταμεία για τους γεωργούς. Ε, Τελευταία ομιλήτρια στον κατάλογο μου είναι η κυρία Μπλεκεβιτσούτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς εδώ συζητούμε κυρίως το θέμα της γεωργίας, έτσι, αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Επέλεξε τον εύκολο τρόπο να τους εντάξει στο Ταμείο Προσαρμογής της Παγκοσμιοποίησης. Το ήξερε όμως ποια αντίδραση θα συναντήσει από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή κρατών μελών. Ωστόσο, επέλεξε τον πιο εύκολο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήθελε ε, τρόπο την να κατευνάσει τους αγρότες και να τους, πείτε, ε, να τους πει ησυχάστε. Θα πάρετε 83% από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχουμε όμως μια κατάσταση τώρα όπου η αγρότες βρίσκονται παγιδευμένοι. Είχε άλλο σκοπό μέχρι τώρα το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχουν βεβαίως το δικαίωμα να υποστηρίζονται οι αγρότες και από το ταμείο αυτό, αλλά εάν πληρούν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους άλλους εργαζομένους, όχι ειδική κατηγορία. Βλέπουμε λοιπόν την αντίδραση των κρατών μελών Άκουσα τις συζητήσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και των κρατών μελών και πολλοί αμφισβητούν πολύ σοβαρά την ίδια την ύπαρξη του Ταμείου αυτού. Εκεί θα πρέπει να συνεργαστεί το Κοινοβούλιο με τα κράτη-μέλη γιατί ακούμε διάφορες απόψεις. Ορισμένα κράτη θέλουν να καταργηθούν τελείως και να έχουμε ένα ταμείο που να υποστηρίζει τους αγρότες μας. Συμφωνώ με τον κύριο Μαν που λέει ότι είναι τα χρήματα περιορισμένα. Ναι. Είναι περιορισμένα και μάλιστα συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη εκεί λόγω και της αλληλεγγύης. Και το Ταμείο αυτό προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση είναι κατεξοχήν Ταμείο Αλληλεγγύης. Ορισμένα κράτη-μέλη ποτέ δεν θα χρειαστεί να προσφύγουν σε αυτό το ταμείο και ελπίζω να μην το χρειαστεί ε, μια χώρα, αλλά άλλες χώρες το χρειάζονται. Η Λιθουανία, ας πούμε, προσέτρεξε αυτό το ταμείο και με επιτυχία αξιοποίησε τα κονδύλια και θέλω να διατηρηθεί η ύπαρξή του και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε εδώ ο κατάλογος λοιπόν. Και ε, θα δώσω λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Λέπρου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένες από τις ερωτήσεις που έγιναν. Πιστεύω ότι ε, βεβαίως υπάρχουν διάφοροι τομείς που θα πρέπει να ε, σκεφτούμε, όχι μόνο τη γεωργία. Ε, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τομείς που να διέρχονται κρίση. Αυτό θα μπορούσε να είναι ως προσέγγιση ενδιαφέρουσα, ε, όσο και καινοτόμα. Και οι συνάδελφοί σας της Επιτροπής, νομίζω, εξωτερικού διεθνούς εμπορίου πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Για τη διετία θα ήθελα να θυμίσω, αν μου επιτρέπετε, ότι το Ταμείο αυτό έχει ως αποστολή να ενισχύει κάποιους εργαζομένους που δυσκολεύονται πάρα πολύ να ξαναβρούν δουλειά. Και αυτό σημαίνει ότι θα διέλθουν μια μακρά περίοδο μετεκπαίδευσης, επανακατάρτισης και μπορεί οι ενισχύσεις να χρειαστεί να καταβάλλονται μια διετία. Σε ό,τι αφορά ε, ξεχωριστή γραμμή στον προπολογισμό, θα ήθελα να θυμίσω ότι ήδη σήμερα, ενώ είμαστε εκτό προπολογισμού, μας προσάπτουν καμιά φορά ότι απορροφούμε μόνο ο κλάσμα των κονδύλιων ε, των διαθέσιμων κονδυλίων. Ας ξεχάσουμε αυτή την προσέγγιση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διαθέσιμα κονδύλια. Παρεβαίνουμε μόνο εφόσον το ζητήσουν τα κράτη-μέλη, διότι έχουν ανάγκες. Και όσο λιγότερο επεμβαίνουν, τόσο καλύτερο. Η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν ε, μηδενική απορρόφηση ουσιαστικά αυτών των πόρων. Αυτό θα σήμαινε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα στη διάθεσή τους για να βοηθήσουν τους εργαζομένους να βρουν δουλειά. Και ότι οι επιχειρήσεις επίσης τους βοηθούν και εμείς δεν χρειαζόμαστε. Τώρα, εάν δημιουργήσουμε ξεχωριστή θέση στον προπολογισμό, κινδυνεύουμε να μας κατηγορήσουν ότι ε, δεν την απορροφάτε αυτή τη γραμμή, τι τη θέλετε. Γιατί όντως τότε θα υπάρχουν κονδύλια ε, που δεν θα απορροφούν. Σας παρακαλώ να έχετε υπόψη σας αυτή την ιδέα ότι πρόκειται για ένα μέσο που έρχεται να αντιμετωπίσει επίγουσες καταστάσεις και ελπίζουμε όσο γίνεται πιο σπάνιες, άρα δεν θα πρέπει να έχει ένα πάγιο τακτικό προπολογισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο για τα κατόφλια και ιδιαίτερα για τους αυτοαπασχολούμενους αντίθετα το γεγονός ότι διευρύνθηκαν οι κατηγορίες ε, επιλέξιμων εργαζομένων και στους ε, ελεύθερους επαγγελματίες και εκείνους που έχουν ε, μια μικρή επιχείρηση ή τη διευθύνουν. Έτσι διευκολύνουμε τη δυνατότητα να βρούμε 500 απολυμμένους ή ε, εξισωμένους, θεωρούμενους ως απολυμμένους. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ανάληψης της επιχείρησης από τους εργαζομένους. Θα μπορούσε αυτό να γίνει ήδη από σήμερα σε περίπτωση που απολύονται οι εργαζόμενοι. Θα μπορούσαμε να του βοηθήσουν να αναλάβουν εκείνη την επιχείρηση, α πούμε με ενίσχυση επενδύσεων. Προβλέπεται αυτό στην πρόταση. Ίσως χρειάζεται να σκεφτούμε γιατί είδους επενδύσεις συζητούμε. Δηλαδή το να εξαγοράζει την επιχείρησή σου είναι ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσαμε να ισχύσουμε. Νομίζω είναι εύκολο κάτι τέτοιο να το θεωρήσουμε. Ε, ως προς τη γεωργία τώρα. Πρέπει να θυμίσουμε και πάλι ότι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι ένα μέσο συμπληρωματικό επιπλέον των εθνικών και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υπάρχουν, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή τα διάφορα μέσα της κοινή γεωργικής πολιτικής και ειδικά της κοινή γεωργικής πολιτικής τα μέσα μπορούν να βοηθήσουν να υπάρξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, να επανέλθει η ανταγωνιστικότητα. Εμείς είμαστε, αν θέλετε, η εσχάτη λύση για να βοηθήσουμε στην περίπτωση της γεωργίας κάποιους αγρότες να προσαρμόσουν την παραγωγή τους, να αλλάξουν την παραγωγή τους, αλλά να παραμείνουν αγρότες. Τελευταία στιγμή δηλαδή επεμβαίνουμε εμείς. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και εδώ είναι η διαφορά με την επιλεξιμότητα. Με απόφαση που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή η Κομισιόν ορίζει το κατά πόσο είναι επιλέξιμος ένας τομέας στην περίοδο αναφοράς και δεν θα πρέπει να περιμένουμε αναγκαστικά 10 χρόνια να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα ένας αγρότης με την τράπεζά του πριν επέμβουμε. Μπορεί να γίνει αυτό πιο γρήγορα. Άλλα στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να συνοδεύσουμε και να πλησιώσουμε την ανασυγκρότηση και τις μεταρρυθμίσεις. Αναφερθήκατε σε πολυεθνικές και άλλες. Θυμίζω ότι δεν έχει λήξει ακόμα η προθεσμία για απάντηση σε ένα, μια πράσινη βίβλο για την ε, αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και τις αλλαγές. Εκεί υπάρχει μια σειρά μηνυμάτων που θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοκιμάσει εντό εισαγωγικών, να βολιδοσκοπήσει τους ενεχομένους, ε, βεβαίω και το Κοινοβούλιο, κοινωνικούς εταίρους και άλλους, για τον τρόπο με τον οποίο ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων. Ποια θα είναι η υποχρέωσή τους, οι υποχρεώσεις τους, ποιες υπηρεσίες και ενισχύσεις μπορούμε να εισαγάγουμε σε επίπεδο κρατών μελών. Δηλαδή και αυτό είναι ένα στοιχείο της συζήτησης. Τέλος, μια σειρά κρατών μελών την περασμένη εβδομάδα ε, δήλωσαν ανοιχτά ότι είναι αντίθετα με τη συνέχιση του ταμείου αυτού, βασιζόμενα στην αρχή της επικουρικότητας, λέγοντας ότι Εντάξει, αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να τα λύνει κάθε χώρα ε, μόνη της στο καταλληλότερο επίπεδο που είναι το εθνικό. Άρα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι περιτεύει ένα ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί σε γενικές γραμμές με την διαπίστωση των κρατών μελών, αλλά δεν καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Βεβαίως θεωρεί ότι κατά πρώτο λόγο θα πρέπει να δρουν τα κράτη-μέλη, αλλά σε περίπτωση σημαντικών αναδιαρθρώσεων, σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή ελεγγύη μπορεί να αποδειχθεί, παράδειγμα και ακριβώς λόγω της παγκοσμιοποίησης, διότι είναι υπέρ των πολλών και κατά ορισμένων λίγων. Και αν το ζητήσουν τα κράτη-μέλη, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσιολογικό να μπορεί να δίνει μια επιπλέον ενίσχυση. Και νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία παραδείγματα ακριβώς σεβασμού της επικουρικότητας, ότι θα πρέπει να έρχεται το αίτημα από τα κράτη-μέλη ως συμπλήρωμα της δικής τους δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος. Για να ολοκληρώσει το λόγο έχει τώρα η συγγήτριά μας κυρία Χάρκιν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις πολύ ενδιαφέρουσες συμβολές τους και για τα επικοδομητικά του σχόλια και από την Κομισιόν να ευχαριστήσω. Να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα που έθεξε η κυρία Μπάουερ και άλλοι το ανέφεραν αυτό, το θέμα του κριτηρίου της ε, εξαίρεσης για λόγω κρίσης. Είπατε ότι κάποια κάτι μέλη δεν το θέλουν αυτό και είναι λογικό να φανταστούμε ότι δεν θα το στηρίξουν ε, ένα ταμείο παγκοσμιοποίησης μετά από το 2014. Και γι' αυτό ίσως να είναι και η τελευταία φορά που ασχολούμαστε με το πώς θα μπορούσαμε να τους πείσουμε να το κάνουν. Ξέρω πως η δανεική κυβέρνηση ήταν ε, ξεκάθαρη στη συζήτηση στο Στρασβούργο ότι θα το εγκαταλείψουν, τελείωσε αυτό, δεν θα επανέλθουν παρόσα, ε, ό,τι μάλλον και να λέει το Κοινοβούλιο. Έπειτα, συμφωνώ ότι, κυρία Λάμπερ, ότι η γεωργική πολιτική πρέπει να μεταρρυθμιστεί και ότι εκείνο το τμήμα θα πρέπει ε, να χρησιμοποιηθεί και ότι χρειάζεται να βρεθεί απάντηση όσον αφορά την κατάλληλη στιγμή. Το μόνο, πρόβλημα, το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το μηχανισμό εκτός του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου, θα είναι ότι θα έχει χωριστή γραμμή ενώ και, και ναι μεν αυτό θα επιταχύνει τη διαδικασία αλλά υπάρχουν άλλα ε, προβλήματα. Κάτι το οποίο όμως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε είναι καταρχήν να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την εφαρμογή και ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε η Κομισιόν αφού θα έχει ε, αξιολογηθεί αρχικά μια αίτηση και δεν χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίε, να υπάρχει δυνατότητα κάποιου είδου ε, αντικαταβολή, προκαταβολή, να κάνω κάποιο ποσοστό, ώστε τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να εφαρμόζουν τα μέτρα, ιδιαίτερα σε περιστάσει όπου τα κρατη δεν έχουν τους πόρους για να το κάνουν αυτό οι ίδιοι, τα ίδια. Πώς ακριβώς το κάνουμε δεν ξέρω, αλλά πάντως θα πρέπει να το διερευνήσουμε και να δούμε αν είναι δυνατόν. Και κύριε Νταρντέν, δεν έχουμε ε, διευκρινίσει τα θέματα αρμοδιοτήτων, αλλά συμφωνώ ότι θα πρέπει να επανέλθουμε ακριβώς στο θέμα ότι η Κομισιόν δεν έβαλε στην άκρη 2,5 δις ε, αντί για 3, αλλά ανέφερε ότι αυτό είναι το όριο που θέλει να προτείνει. Οπότε δεν θα απομακρυνθεί καμιά επιτροπή από τα 2,5. Και η μικρή απορρόφηση του Ταμείου επίσης αυτό οφείλεται εν μέρη στο ότι τα κάτι μέλη τώρα άρχισαν να το χρησιμοποιήσουν και πιστεύω ότι θα υπήρχαν περισσότερα αιτήματα και όπως είπε η Κομισιόν ε, η ιδανική κατάσταση θα ήταν να μην χρειάζονται, να μην έχουμε μηδενικές αιτήσει, αλλά ξέρουμε πως αυτό δεν πρέπει να συμβεί σύντομα λόγω της κατάστασης. Πιστεύω πως τα κράτη-μέλη να ε, δεν έχουν ακριβώς δει το άρθρο 4.2 για τα κριτήρια παρέμβαση, ιδιαίτερα τα μικρά κράτη-μέλη, ότι θα μπορούσαν δηλαδή να ζητήσουν σε περιφερειακό επίπεδο χρήματα χωρίς ε, συγκεκριμένη χρονική περίοδο και και πολλά. Κύριε Τόμας Μαν, συμφωνώ ότι δεν μπορεί να κατευθυνθεί προ την Γεωργία, όμω εκεί λέμε για 2,5 εκατομμύρια αντί για 3 για τον προπολογισμό και την εφαρμογή του. Και αυτό είναι η καρδιά πολλών προβλημάτων. Λέτε για τα κράτη-μέλη, ξέρετε ότι υπάρχει το θέμα της ε, μειονότητας ε, που μπλοκάρει το θέμα, ακόμα και αν πολλοί από αυτά τα κράτη-μέλη που είναι εναντίον χρησιμοποίησαν αυτή τη διευκόλυνση πέρυσι. Η κυρία Μπέρες μίλησε για εμπορικές συμφωνίες και νομίζω πως όλοι συμφωνούμε με τα αυτά που είπε και το σχόλιο ίσως για την, ε, κάποιον ε, εργαζόμενοι, αν θα μπορούσαμε δηλαδή να το ξαναεξετάσουμε. Τελειώνω, ναι, δύο λεπτά. Μιλήσατε για προβλήματα πολιτικής ανταγωνισμού. Εγώ θα ήθελα αυτό να το διευκρινίσουμε κάπως περισσότερο, να το συζητήσουμε. Δεν είμαι βεβαία για το ποια είναι ακριβώ τα θέματα και για την πολιτική μετεγκατάσταση. Κύριε Μπένιον, Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι επειδή η Κομισιόν θα το εξετάσει με πράξεις εξουσιοδότηση, μπορεί και να αντιμετωπιστούν κάποια από τα προβλήματα που αναφέρατε. Και κάποιοι που είπαν ότι θεωρούν ότι στο Συμβούλιο η αντίσταση θα είναι μεγαλύτερη αν συμπεριλάβουμε και τους γεωργούς. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό τι θα γίνει. Και κυρία Ζούμπερ, εγώ συμφωνώ μαζί σας για τη συγχρηματοδότηση, αλλά και πάλι αν γινόταν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ε, ταμείο θα έπρεπε να γίνει μέσα στο σημερινό πλαίσιο. Κυρία Μπλίνκεβιτσούτε, έχετε δίκιο ότι θα πρέπει να γίνει σύντομα αυτή η υπόθεση να δώσουμε κάποια ποσά. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με όλα αυτά στην Επιτροπή μας και ε, προσπαθούμε να χειριστούμε ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Τέλος, εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε το Ταμείο η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει με τις τροπολογίες της και με τις προτάσεις της ότι, την απόδειξη της χρησιμότητας και το τελικό μου σχόλιο για το ότι προσπαθούμε να πείσουμε ορισμένα κάτι μέλη ότι το χρειαζόμαστε και είναι καλή ιδέα. Ένας τρόπος ήταν να δούμε τις επιλέξιμες δράσεις και αυτές να τις ε, συνδέσουμε με την πραγματικότητα, γιατί αφού έχω μιλήσει με εργαζόμενους που επωφελήθηκαν από το ταμείο αυτό και φαντάζομαι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει το ίδιο, σίγουρα σε κάποια κάτι μέλη, πιστεύουν λοιπόν πως πολλές από τις παρεμβάσεις θα είχαν γίνει ούτως ή άλλως από τις εθνικές κυβερνήσεις και θέλουν να δουν προστιθέμενη αξία. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν αυτό να το χρησιμοποιήσουμε ως επιχείρημα, να είναι πια ορατή η προστιθέμενη αξία για τις δράσεις που γίνονται και ίσως και κάποια ευθυγράμμιση για το κάποια αν είναι στόχοι της Ευρώπης 2020, εθνική στόχη με άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως αυτό θα μπορούσε να πείσει τα κράτη-μέλη πως το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση έχει αξία. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Την εισηγήτρια. Σε εκείνη τώρα να πόκειται και να λύσει το πρόβλημα. Γιατί μόνο αν βρει εκείνη κάποια λύση θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να δούμε και ποια θα είναι τα χρονοδιαγράμματα. Γι' αυτό δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω τίποτα για προθεσμίες. Τις επόμενες μέρες μάλλον θα αποφασιστούν διάφορα πράγματα και θα σας ενημερώσει η γραμματεία όλους σας. Μπορώ λοιπόν εδώ να κλείσω τη συνεδρία. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 9. Καλό σας βράδυ.